για να ασκήσει πίεση και να έρθει πιο πολύ κοντά στις δικές μας απόψεις. Ευχαριστούμε. Έκλεισε λοιπόν η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Τώρα, περνάμε στην δήλωση της Αντιπροέδρου ε, της ε, Επιτροπής ε, σχετικά με το γενετικό ακροτηριασμό εκ μέρους λοιπόν της κυρίας Άστον. Θα λάβει το λόγο ο Επίτροπος κύριος Ντάλι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάθε είδους βίας με βάση το φύλλο ε, συνιστά απαράδεκτη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ε, μεγάλο ε, εμπόδιο για την ισότητα των φύλων. Ο εκροτηριασμός των γενετικών οργάνων των γυναικών είναι ένα είδος βίας κατά των γυναικών που είναι ιδιαίτερα απαράδεκτη και ιδεχθής. Είναι υποτιμητικό, παραβιάζει ουσιαστικά θεμελιώδη δικαιώματα και το δικαίωμα το ίδιο στην υγεία και δικαιώματα των παιδιών όλος ιδιαίτερος. Τρία εκατομμύρια εκτιμάται ότι είναι οι γυναίκες και τα κορίτσια στον κόσμο που κάθε χρόνο υφίσταται ε, ακροτηριασμό ε, των γεννητικών τους οργάνων. Περίπου μισό εκατομμύριο γυναικών που ζουν στην Ευρώπη ήδη το έχουν υποστεί και πολλές χιλιάδες ακόμα κινδυνεύουν. Ε, ακροτηριασμός των γυναικείων ε, γεννητικών οργάνων δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση για λόγους παραδοσιακούς, πολιτιστικούς και πρακτικές αιώνων. Έχει επιπτώσεις και άμεσες και μακροπρόθεσμες στην υγεία των γυναικών και μπορεί να προκαλέσει μέχρι και το θάνατο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να αναλάβει συγκεκριμένη δράση και πολιτική να απαντήσει στεναρά για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα της βίας κατά των γυναικών στην Ευρώπη. Ο ακροτηριασμό των γυναικείων ε, γεννητικών οργάνων ε, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο. Έχουμε μια στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ισότητα ανδρών και γυναικών πενταετούς διάρκειας 2010-2015. Δεν έχουμε αξιόπιστα στοιχεία και συγκρίσιμα. Είναι τεράστια πρόκληση αυτό. Ο συνάδελφός μου αντιπρόεδρος κυρία Βιβιάν Ρέντινγκ ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ισότητας των Φύλων να εκτιμήσει την αξιοπιστία και την διαθεσιμότητα των ε, δεδομένων και των στατιστικών στοιχείων από τα κράτη-μέλη και να εντοπίσει τις ελλείψεις. Αυτό λοιπόν το Ινστιτούτο θα ε, κάνει μια καταγραφή της κατάστασης και θα απαντήσει τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Αναμένεται η έκθεση στο δεύτερο ήμιση του ε, ενεστώτος έτου. Το αποτέλεσμα αυτό θα μας βοηθήσει βοηθήσει να λάβουμε καλύτερα μέτρα με τα λόγου γνώσεως. Το 2011-2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε και κονδύλια για την καταπολέμηση τέτοιων βλαβερών ε, πρακτικών. Οικονομική ενίσχυση θα δοθεί για διεθνή προγράμματα, για οργανώσεις που δρούν επιτόπου και εργάζονται για την πρόληψη τέτοιων πρακτικών με αύξηση της συνειδητοποίησης και με αλλαγή κοινωνικών συμπεριφορών παρόλο που δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία για το θέμα αυτό ε, ε, είναι ποινικό αδίκημα στα περισσότερα κράτη-μέλη είτε με ειδικού νόμους διώκεται ή στο Γενικό Ποινικό Κώδικα. Μια μεγάλη πλειοψηφία κρατών μελών της Ένωσης έχει περιλάβει την ίδια την αρχή ε, της ετεροδικίας στο ποινικό τους κώδικα και έτσι μπορούν να διώκονται ε, αδικήματα αξιόπινης πράξης ακροτηριασμού που έχουν ε, τελεστεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ποινική δικαιοσύνη προτείνουμε μέτρα και νομοθεσία ε, για τα δικαιώματα των θυμάτων ε, εγκληματικών πράξεων. Με την οδηγία για τα θύματα στοχεύουμε στην προστασία των θυμάτων παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έχουν κάποια βασικά ελάχιστα δικαιώματα και να αντιμετωπίζονται ως άτομα, ως πρόσωπα ε, ξεχωριστά ε, το κάθε θύμα και να έχουν την αντίστοιχη θεραπεία. Οι ανάγκε των θυμάτων θα πρέπει να εκτιμώνται σε ατομική βάση και τα πιο ευάλωτα πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων ε, ε, του ακροτηριασμού των γυναικείων ε, γεννητικών οργάνων να τη χάνουν της ανάλογης αντιμετώπισης και θεραπεία. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τι αλλαγέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βελτιώσει ουσιαστικά την κατάσταση των γυναικών που είναι θύματα βία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης αντιμετωπίζει αυτό το θέμα του ακροτηριασμού των ε, γεννητικών οργάνων των γυναικών στην εξωτερική δράση. Ε, υποστηρίζει ε, δραστηριότητες λόμπι και προστασίας και δικαστική και νομικής για να αποτραπούν τέτοια φαινόματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση συστηματικά θέτει αυτό το ζήτημα στο διάλογο με χώρε Αφρική, Καραβική και Ειρηνικού. Και σε αυτό το πλαίσιο υπογραμμίζουμε την ανάγκη οι αφρικανικές χώρες να βεβαιώνουν ότι απαγορεύεται στις χώρες του ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και να εφαρμόζεται αυτή η απαγόρευση. Υποστηρίζουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο ψήφισμα που σχεδιάζει για να απαγορεύσει ε, αυτή την πρακτική. Είναι, είναι κρίσιμο οι χώρες όπου απαντάται περισσότερο αυτό το φαινόμενο που είναι χώρε αφρικανικές ιδίω, να κάνουν κτήμα τους ε, και να εφαρμόσουν αυτό το ψήφισμα. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ένωσης αυτό τον καιρό προετοιμάζει εκστρατεία ε, υπό τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών για να επιστήσει την προσοχή στην ανάγκη να ε, ενταθούν οι προσπάθειες για να εκριζωθεί αυτή η πρακτική ιδιαίτερα από την Αφρική. Ε, ο κριτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι ακραία πρακτική και απαράδεκτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να την καταπολεμήσει και να βοηθήσει τις γυναίκες και να ε, τις ενδυναμώσει και στην Ένωση και εκτός της ε, Ένωσης με νομοθεσία, οικονομικά μέτρα και μια σειρά άλλων μέσων και μεταξύ αυτών υποστήριξη οργανώσεων επιτόπου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Επίτροπε, τώρα θα ακούσουμε τους ομιλητές από πλευράς των πολιτικών ομάδων και αρχίζουμε με την κυρία Μουσκαρδίνη από πλευράς του Έλκα για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κροτηριασμός των ε, γεννητικών οργάνων και η καταπολέμηση αυτού είναι ένας διαρκής ε, αγώνας. Ε, πρόκειται για μια μάστιγα που επηρεάζει τις γυναίκες για ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή τους. Θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτή η ποινική πράξη με τις ίδιες κυρώσεις, με τα ίδια δρακόντια μέτρα που προβλέπονται για άλλα δικήματα. Τελικά αναγνωρίστηκε ότι πρόκειται για κατάχρηση το για παραβίαση μάλλον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών ε, όταν ε, τους ακροτηριάζουν τα γενετικά όργανα και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το θάρρος αυτών των γυναικών που παρά τις απειλές ε, από την περιβάλλουσα κοινωνία συνέχισαν τον αγώνα τους για την καταπολέμηση αυτής της πρακτικής. Είναι πάρα πολύ Σημαντικός ο ρόλος αυτών των γυναικών, ε, ε, αυτό το φαινόμενο παρατηρείται και σε διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και οι παραδόσεις, οι φιλετικές αυτές παραδόσεις συνεχίζονται. Θα πρέπει να απαγορευτεί αυτή η αξιόπινη πράξη και γι' αυτό μέσα στα σημεία 6, 7 και 8 ζητούμε δράση άμεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταπολεμηθεί αυτή η μάστιγα, η στρατηγική καταπολέμηση στη βίας κατά των ε, γυναικών πρέπει να συνεχιστεί. Υπάρχουν εκστρατείε ενημερωτικέ για τον ακροτηρισμό των γεννητικών οργάνων, παραδείγματο χάρη ενημερωτικέ εκστρατείε για νεαρά κορίτσια και εντό και εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω αναφέρουμε στο ψήφισμά μα, σχετικά με τον ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων και παρόδο να σημειώσετε ότι το Φεβράριο του 2009 έχει εγκριθεί με συντριπτική πλειοψηφία αυτό το ψήφισμα. Υπάρχουν ε, λοιπόν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σε αυτό το ψήφισμα. Παρόλα αυτά που μα είπε όμω ο Επίτροπο Ντελή σήμερα, Νταλή, σήμερα δεν ε, ε, επαρκεί η δράση μα και αυτό το ποινικό αδίκημα δεν αντιμετωπίζεται Όπω άλλα παρεμφέρει. σα ευχαριστούμε. Η κυρία Γκόμε, τώρα ε, από πλευρά των σοσιαλιστών. Ο ακροτηριασμό ε, των γεννητικών οργάνων των γυναικών δείχνει την ανισότητα των δύο φύλων. Πρόκειται για βία κατά των γυναικών, κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών και δεν αιτιολογείται με οποιοδήποτε επιχείρημα και αν προτάξουμε η καταπολέμηση της βίας ε, κατά των γυναικών πρέπει να συνεχιστεί στα πλαίσια του γενικότερου αγώνα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη και οι εταίροι θα πρέπει να συντονίζουν τη δράση τους ώστε να είναι ρηξικέλευτα τα προγράμματα που θα καταπολεμήσουν αυτές τις πρακτικές, να βοηθήσουμε αυτά τα νεαρά κορίτσια που βρίσκονται σε τόσο ευάλωτη θέση, να τους προσφέρουμε υπηρεσίες και προγράμματα ενημέρωση. Επίσης, η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συνεχίσει τα προγράμματα προγράμματά τη να συνεχίσουμε την κινητοποίηση και την ευαισθητοποίηση ε, που βοηθούν ε, τις πληθυσμιακέ ε, ομάδε που βρίσκονται σε κίνδυνα εντό και εκτός τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Θα ακολουθηθούν λοιπόν οι συστάσει του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόσο ώστε τα δικαιώματα των γυναικών και η χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών να ενταχθούν σε, σε τι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση, Ένωσης για την ισότητα των δύο φύλων. Οι εθνικέ περιφερειακέ και τοπικέ αρχέ, η κοινωνία των πολιτών σε τρίτε χώρε, όλοι μαζί πρέπει να συνεργαστούν συνεργαστούμε για να το πολεμηθεί το φαινόμενο. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρου των ε, φιλελευθέρων Μπιλμπάου. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Μάστιγα είναι ο κροτηριασμός γεννητικών οργάνων των γυναικών και είναι κατάφορη ε, δήλωση ε, διαφοράς των φύλων. Σε κάποιους πολιτισμούς οι γυναίκες είναι κτήματα των ανδρών και με τη βία τους επιβάλλουν την δεσμόζουσα θέση τους, την κυρίαρχη θέση τους και κάποιους μύθους και εικασίες. Οι άνδρες δικαιολογούν και όλα σε αυτή την πρακτική ε, θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στα θύματα. Όλες οι γυναίκες στον κόσμο θα πρέπει να μάθουν ότι ο ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων είναι απαράδεκτος για λόγους αξιοπρέπειας. Και ε, οι άνδρες θα πρέπει να μάθουν ότι οι ανασφάλειες και οι φόβοι τους ε, θα πρέπει να καταρριφθούν. Ε, το φαινόμενο αυτό χρειάζεται ενιαία αντιμετώπιση με ευρωπαϊκό κανονισμό και με ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης για να εκκριζωθεί το φαινόμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από τους Πρασίνους η κυρία Ντουιράν παρακαλώ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι κάτι που υποστηρίζω το ψήφισμα και ελπίζω αύριο να το ψηφίσουμε ομόφωνα γιατί είναι τόσο προφανές και αυτονόητο και εγγράφεται σε μια στρατηγική ε, διεθνή στρατηγική για την ε, απαγόρευση των γεννητικών ακροτηριασμών σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Και είναι πολύ σημαντικό με το δικό μας ψήφισμα να υποστηρίξουμε τη διεθνή στρατηγική. Πολλές γυναίκες ε, είναι εκεί δεσμευμένες. Η κυρία Σαντάλ Κανταωρέ, η πρώτη κυρία της Μπουρκίνα Φάσο, για να γίνει διεθνής προσπάθεια και άλλες γυναίκες και άλλες χώρες προσυπογράφουν αυτή την απαγόρευση. Θα πρέπει να προωθήσουμε αυτό το θέμα. Μπορεί να συνεισφέρει στη Γενική Συνέλευση του ε, το δικό μας ψήφισμα και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η απαγόρευση είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα και πολιτικό μήνυμα αλλά δεν μας απαλλάσσει από το να εργαστούμε ε, παντού με ομάδες γυναικών, με γυναίκες που κάνουν αυτές τις πρακτικές γιατί δεν είναι πάντα άντρες. Όχι, σχεδόν ποτέ δυστυχώ γυναίκες τις κάνουν αυτές τις ε, επεμβάσεις και θα πρέπει να υποστηριχθούμε αν υπάρχει γενικευμένη απαγόρευση από τον ΟΗΕ, όπως και για άλλα θέματα της νάρκες κατά προσωπικού, θα ακολουθήσει η στρατηγική με παρακολούθηση ε, και είναι πολύ σημαντικό θέλουμε τελικά να εκκριζωθεί αυτή η μάστιγα για όλες τις γυναίκες του κόσμου. Ευχαριστώ. E Εκ μέρου των Ευρωπαίων Συντηρητικών Μεταρρυθμιστών, κύριε Γιανακουδάκη, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, ντρέπομαι που πρέπει να πω ότι ο αριθμός ε, των περιπτώσεων γεννητικών ακροτηριασμών στην δική μου εκλογική περιφέρεια στο Λονδίνο αυξάνεται ορισμένες από αυτές τις διαδικασίες μάλιστα γίνονται στο ίδιο το Λονδίνο γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι που σήμερα έχουμε αυτή τη συζήτηση ε, διότι ο ακροτηριασμός αυτός γίνεται σε γυναίκες που ζουν στην Ευρώπη ο ακροτηριασμός είναι νόμιμος ε, ε, στην Ευρώπη και μπορεί να γίνει αυτό ακόμα και αν οι γυναίκες μεταφέρονται στο εξωτερικό. Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, καταπολεμήσουν στεναρά αυτή την παράνομη πρακτική. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να προστατεύσει τις νέες κοπέλες και τις γυναίκες και να δώσει το καλό παράδειγμα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ο κροτηριασμός είναι βάρβαρος, αποτελεί κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων δικαιωμάτων των γυναικών και των νέων κοριτσιών. Είναι θέμα ταμπού. Ελπίζω λοιπόν ε, μιλώντας ε, για το θέμα αυτό ανοιχτά ε, θα μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε αυτή την ολέθρια πρακτική. Πολύ ωραία για την εκμέρωση της ο κύριος Γκούσταψον για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι όπως και οι συναδελφοί μου ε, που θα εγκρίνουμε αυτό το κοινό ψήφισμα το οποίο στηρίζει τις εργασίες ε, των Ηνωμένων Εθνών και διαπιστώνει ότι εδώ πρόκειται για απαράδεκτες ε, πρακτικές. Θέλω να πω ότι η αγώνας κατά της, του γενετικού ακροτηριασμού πρέπει να συμβαδίζει με την καλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Το θέμα είναι το εξής. Ε, τα σεξουαλικά και αναπαγωγικά δικαιώματα των ε, γυναικών πρέπει να προστατευτούν. Ε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να επιλέγουμε κάποιους πολιτισμούς αφορά το θέμα όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια. Όμως παράλληλα είναι σημαντικό να συνεργαζόμαστε με οργανώσεις ε, γυναικών και άλλους αρμόδιους φορείς. Παρακαλούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει μια πρόταση για μια ευρωπαϊκή στρατηγική γιατί μόνο με τέτοια στρατηγική θα είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τον γενετικό ακροτηριασμό των γυναικών στην Ευρώπη. Η κυρία Ματέρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε ε, θέλω να πω με απόλυτη πειθό είμαι ακράδαντα πεπισμένη ότι είμαι υπέρ αυτού του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αντιμετωπιστεί αυτή η βάρβαρη πρακτική ε, του ε, γενετικού ακροτηριασμού. Είναι απάνθρωπο αυτό που συμβαίνει και αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο πρέπει να αντισταθούμε σε μία πράξη που ε, αφορά πάρα πολλές γυναίκες, περίπου 500.000 μόνο στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τη διακριτική μεταχείριση ε, την οποία υφίσταται το γυναικείο φύλλο. Οι γενετικοί ακροτηριασμοί προκαλούν ε, αμετάκλητες συνέπειες ε, για την φυσική κατάσταση της γυναίκας. Μολύνσεις, κίνδυνος προσβολής από το AIDS, συνέπειες στους τοκετούς. Αυτά είναι μόνο κάποια από τα, κάποιες από τις συνέπειες που προκαλούνται από αυτές τις ε, πρωτόγονες ε, πρακτικές χωρίς αποστήριση αποστήρωση. Ε, αυτό γίνεται και σε γυναίκες κάτω των 15 ετών. Ε, εδώ μιλώ, μιλάμε λοιπόν για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως των δικαιωμάτων των παιδιών. Είναι λοιπόν απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει αυτό το έγκλημα έτσι ώστε να διοχετεύσει τα απαραίτητα κονδύλια για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Και είναι απαραίτητο να στηρίξει την πράξη αυτή το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού αυτή την ε, συνεχιζόμενη βία που ασκείται σε όλες τις γυναίκες του κόσμου. Ευχαριστούμε πολύ. Kaiser για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ποτίσω φόρο τιμή σε όλα τα κορίτσια, σε όλε τι γυναίκε που έχουν ακροτηριαστεί. Ε, γιατί έχουν υποφέρει. Πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό ο ακροτηριασμό. Νομίζουμε όλοι ότι περικόπτεται μόνο η κλητορίδα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ε, είναι επίσης ότι αφαιρούνται τα χείλη του εδίου και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται από δέντρα βελόνες για να ξαναραφθεί ε, ο κόλπος ο οποίος καλύπτεται στη συνέχεια και ε, για να επιτραπεί η ούρηση εισάγεται σε μία μικρή οπή ένα καλάμι για να περνούν και οι διάφορες γεννητικές εκκρίσεις. Μόνο και μόνο για να ορίσει η γυναίκα χρειάζεται μία ώρα και στη συνέχεια όταν θα έχουν περίοδο αυτά τα κορίτσια πρέπει να εισαγάγουν ένα νέο καλάμι μέσα στον κόλπο ε, και ε, ε, κυλιούνται ε, από τον πόνο κάτω στο πάτωμα ε, τα κορίτσια και έχω συναντηθεί με γυναικολόγους στις Βρυξέλλες ε, που ανακάλυψαν γυναίκες που γεννούσαν ενώ υπήρχε αυτό το καλάμι και δεν επέτρεπαν την αφαίρεσή του οι γιατροί. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτός ο ακροτηριασμός πρόκειται για μια χιλιετή παράδοση που υπήρχε ακόμη και στη χριστιανική χριστιανική παράδοση με την ζώνη της αχνότητας ε, που έφεραν οι γυναίκες παραδείγματος χάρη των σταυροφόρων. Ε, πρόκειται λοιπόν ε, για τον ίδιο αγώνα όλων των γυναικών ανά τον κόσμο για την ελευθερία τους. Πρόκειται για ένα σκοταδισμό της θρησκείας που διονύζει μπροστά στα μάτια μας σε αυτό το βασανιστήριο. Πρέπει να σταματήσει αυτή η πρακτική και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει άμεσα δράση. Σας ευχαριστούμε τώρα η κυρία Βίξτρομ ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο ακρατορισμός ε, των ε, γενετικών οργάνων είναι κάτι το περίγραπτο. Δεν βρίσκω τις λέξεις. Τρία εκατομμύρια γυναίκες το χρόνο υποφέρουν από αυτό. 8.000 τη μέρα δηλαδή. 240 γυναίκες την ώρα ή 5 γυναίκες το λεπτό που υφίστανται αυτή την μεταχείριση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοηθήκανε πόσο μεγάλο είναι ο πόνος. Ε, αφήστε τα στατιστικά στοιχεία. 180.000 κορίτσια στην Ευρώπη βάσει των πληροφοριών βρίσκονται σε ζώνη κινδύνου και ε, κινδυνεύουν από αυτή την βάρβαρη πράξη. Τώρα ε, υπάρχουν κινήσει για μια παγκόσμια απαγόρευση του ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων. Θα πρέπει αυτό να αναδειχθεί σε ύψιστη προτεραιότητα στα πλαίσια του αγώνα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε συνδυασμό με αυτό το ψήφισμα ε, γιατί είμαστε πολλοί που προσυπογράψαμε και το θεατρικό έργο ε, «Ο μονόλογος ε, του κόλπου», «Vagina Monologue», που επέκτηκε στο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πέραν κάθε ιδεολογίας, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να σταματήσει αμέσως αυτή η βαρβαρότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα, Κιλ Νίλσεν, για ένα λεπτό. Θα σας μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία σε αυτό το θέμα. Στη συνεργασία την αποκεντρωμένη είχα την ευκαιρία να εργαστώ στην Αφρική και να δω ε, τι εστί ο ακροατηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων που ανέφερε η κυρία Ντεκεζέ. Το ψήφισμά μας επιμένει να βασιστούμε στις τοπικές αρχές και τις ΜΚΟ. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρακτική. Σε κάθε ε, είδους καταπολέμηση του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι γυναίκες θα κάνουν αυτά και είναι επαγγελματίε ε, και είναι το μοναδικό του εισόδημα πολλές φορές αυτή η δραστηριότητα και ξέρω ότι πολλές από τις γυναίκες αυτές είναι πρόθυμες να εγκαταλείψουν την πρακτική αν τους προτείνει κάποιος επαγγελματική επανένταξη. Θα ήθελα πραγματικά να σας αναφέρω την προσωπική προσωπική μου εμπειρία. Το έχω ζήσει. Επίσης θα ήθελα να επιμείνω ε, στον υποδειγματικό χαρακτήρα των αντιπροσωπιών που στέλνουμε στις τρίτες χώρες και θα πρέπει να είναι ισομερείς. Γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος να μεταφέρουμε την ισότητα ανδρών και γυναικών. Grazie la parola all'onorevole McClarkin per un minuto. McClarkin, για ένα λεπτό. Κύριε Ως νέα διάβασα με τρόμο μια ιστορία ε, μιας ε, άμεσα ενδιαφερόμενης. Δεν το έχω ξαναδιαβάσει στο παρελθόν και δεν ήξερα καν τι ήταν. Έδειξε το, το μυρό ε, τόλμη θάρρος και ε, μίλησε για αυτά τα πράγματα η γυναίκα αυτή. Αξίζει το θαυμασμό μας και δείχνει ότι εκατομμύρια γυναικών σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από αυτά τα ε, τρομερά και την πρακτική αυτή. Δυστυχώς ο κροτηριασμός των γυναικείων οργάνων ε, δεν είναι άγνωστο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράνομα 100.000 ε, γυναίκες υφίστανται αυτή την πρακτική και κορίτσια μέχρι και 10 ετών. Είναι βαρβαρότητα αυτή η δραστηριότητα. Και δεν είναι μόνο ε, σωματική βλάβη αλλά και ψυχική για όλη τους τη ζωή. Αυτό ε, θα πρέπει να το πούμε είναι ανίποτα τα δεινά τους. Και δεν είναι μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού παραβιάζονται. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εκριζωθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη και παντού αυτή η βάρβαρη πρακτική και αυτό το ιδεχθές έγκλημα. Ευχαριστώ κυρία Πιετικάινεν. Ένα μισή λεπτό. Τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να γίνουν σεβαστά σε όλους τους τομείς της ζωής με τη δέουσα νομική ε, ασφάλεια. Δεν σχετίζεται αυτό με προσωπικά ιδανικά είναι καθολικά, οικουμενικά ε, δικαιώματα, δικαιώματα που έχει κάθε γυναίκα, κάθε κορίτσι, κάθε παιδί. Και δεν μπορούν να ε, υπαχθούν στην αρχή της επικουρικότητας. Δεν είναι δουλειά των κρατών μελών ή οποιονδήποτε κρατών ε, να αποφασίσουν για το πώς μεταχειρίζονται το ίμιση του πληθυσμού τους μία από τις πλέον και βάρβαρες δράσεις είναι ακριβώς ο ακροτηριασμός των γεννητικών οργάνων διότι αυτό σχετίζεται με τον ε, πυρήνα της ε, προσωπικής ε, ταυτότητας του φίλου ενός ανθρώπου. Με τον ακροτηριασμό αυτό ακροτηριάζεται ολόκληρη η γυναίκα ε, διότι αναιρείται η σεξουαλική της ε, ύπαρξη, η αναπαραγωγική της υγεία, ολόκληρη της ύπαρξη. Ε, οι γυναίκες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για την τύχη του σώματος και του πνεύματος τους, να κάνουν τις επιλογές για τη ζωή τους, ανεξαρτήτως προτιμήσεων. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δράσουν το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τα κράτη μελη στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στο πολυμερές επίπεδο, δηλαδή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα πρέπει να κινηθούμε εν ώψη της επικείμενης Γενικής 67ης Γενικής Συνέλευσης, ώστε να εγκριθεί το ψήφισμα για να απογορευτεί παγκοσμίω ο ακροτηρισμό των γεννητικών οργάνων των γυναικών. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Γιγιόμ τώρα για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα με τη σειρά μου ε, να ζητήσω να θέσουμε να πέρα ε, σε αυτό ε, το φαινόμενο του ακροτηριασμού. Δεν πρέπει να ξεχνούμε αυτά που συμβαίνουν ε, στον ΟΗΕ, ε, τα τεκτενόμενα στα κράτη-μέλη και θα σχολιάσω ένα συγκεκριμένο στοιχείο που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Εκτιμάται ότι 180.000 γυναίκες εκτίθενται σε σοβαρό κίνδυνο και δέχονται διώξεις λόγω φύλου και θρησκείας και βάσει πρόσφατης νομολογίας αποδεικνύεται ότι εάν κάποια γυναίκα ζητήσει άσυλο διότι κινδυνεύει να υποστεί ε, τον ακροτηριασμό ε, ή τον έχει ήδη υποστεί βάσει του άρθρου 51 δικαιούται την χορήγηση ε, του ασύλου. Τα κράτη-μέλη όμως ερμηνεύουν περιοριστικά τα κριτήρια για την χορήγηση αυτού του καθεστώτος. Δεν πρέπει όμως να επιτρέψουμε αυτόν τον κατακαιρματισμό διότι χρειάζεται να δράσουμε όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα για να καταπολύσουμε καταπολεμήσουμε αυτό το αδίκημα που ακόμη δεν τιμωρείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ε, ε Χιμένες τώρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τότε που μπήκα στο κοινοβούλιο δεν σταμάτησα να καταγγελώ τον ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Είναι ασιοπηρό έγκλημα και το δέχονται και το υποφέρουν 70 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω, 70 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια. Είναι απαράδεκτο, αφόρητο αυτό το νούμερο και συνέπειες τεράστιες. Έχουμε ψυχολογικές συνέπειες, υγείας, θρησκευτικές προφάσεις όλα αυτά. σε κορίτσια το κάνω, σε ηλικίε μικρές και 14 ετών και κάτω μέχρι και ενό έτου. Ε, και είναι βαριά ε, τα τραύματα, όχι μόνο σωματικά και ψυχικά. Θα πρέπει με όλες μας τις δυνάμεις να εκριζώσουμε αυτή την πρακτική. Ε, δεν υπάρχει ισότητα ανθρώπων και γυναικών, ισότητα ευκαιριών. Απειλείται η ζωή, είναι κακομεταχείριση, βαρβαρότητα, βασανιστήριο. Τι να πω κατά των κοριτσιών. Και αυτό ε, μεταναστεύει και στην Ευρώπη. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε όλους τους μηχανισμούς πρόληψης που έχουμε στο νομικό μας σύστημα και καλό τους ε, δικαστές να ε, προλάβουν αυτό το φαινόμενο να τιμωρούν εκείνους που κάνουν αυτές τις πρακτικές. Η φωνή της Ευρώπης να είναι μία ως προς τον νόμο και ζητώ από την κοινωνία των πολιτών και τις ΜΚΟ να συμπεριληφθούν ε, ενεργά εκστρατείε πρόληψης και ενημέρωσης. Βεβαίως έχουμε πολύ δρόμο, αλλά είμαστε πολλές και πολλοί και δεν θα σταματήσουμε γιατί το οφείλουμε σε 70 εκατομμύρια επαναλαμβάνω γυναικών και κοριτσιών που έχουν υποστεί ακροτηριασμό. Πολύ ωραία. Κάσμαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, εγώ θα συμφωνήσω με όλα αυτά που ήδη ελέγχθησαν. Ο αγκτηριασμός ε, είναι ε, μια κατάχρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των παιδιού και των γυναικών ε, σε όλο τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε αυτά τα ολιστικά δικαιώματα των γυναικών. Ε, και εδώ περιλαμβάνονται και η σεξουαλική υγεία και το δικαίωμα αναπαραγωγή. Το δικαίωμα τη γυναίκα να αποφασίζει μόνη τη τι θα κάνει με το σώμα τη. Κυρία Πρόεδρε, και εγώ ήμουν μάρτυρα των φυσικών συνεπειών σε γυναίκε που εξαναγκάστηκαν να υποστούν αυτό τον γεννητικό και αυτό είναι φρικαλαίο, είναι βάρβαρο. Κανένας πολιτισμός, καμία θρησκεία δεν μπορεί να υπεραμείνεται αυτού. Ε, η συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κατά την 67η Σύνοδό της θα εξετάσει αυτό το τόσο σημαντικό θέμα και χαίρομαι που η ομάδα της Αφρικής ε, και αυτή θα επιληφθεί του θέματος. Αυτά όμως ε, συμβαίνουν όχι μόνο και στην Αφρική και σε άλλες υπηρεσίες αλλά όπως ελέγχεται προηγουμένως και εδώ στην Ευρώπη. Μιλάμε, Μιλάμε για 500.000 γυναίκες που ζουν με τις συνέπειες ε, του ανκτηριασμού και 180.000 εξακολουθούν να κινδυνεύουν. Μην ξεχνάτε λοιπόν αυτές τις 180.000 γυναίκες ε, και τα νέα κορίτσια που κινδυνεύουν. Είναι ντροπή για όλους μας. Grazie. Ora darò la parola agli oratori che l'hanno chiesta con il catch di Sono però ε, έχουν ζητήσει πάρα πολύ το λόγο στο πλαίσιο του Catch the Eye. Ε, θα ήθελα όμως ε, να σκεφτείτε το ένα λεπτό. ξεκινάμε με κόρκολα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πέρσι είχαμε καλές ειδήσει, ε, καλά νέα όταν έγινε η εκστρατεία του ΟΗΕ για αυτό το θέμα και έτυχε μεγάλη υποστήριξη. Βεβαίως οι δεχθεί πράγματα συνεχίζουν να συμβαίνουν Δυστυχώ. Ο ακροτηριασμό των γενετικών οργάνων αποτελεί μια ευρύτατα διαδεδομένη πρακτική διότι αντιλαμβάνεστε ότι σε κάποια μέρη του κόσμου πάνω από το 70 ή το 80% του γυναικείου πληθυσμού ε, εκτίθεται σε αυτόν τον κίνδυνο. Η πρακτική πρέπει να σταματήσει μόνο και μόνο για λόγους υγείας. Ε, ε, είναι ένα μείζον πρόβλημα και θα πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο ούτω ώστε να πάψει αυτή η πρακτική είτε βασίζεται στην θρησκεία είτε όχι. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου και να ε, οργανώσουμε εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι πρόκειται για ένα έγκλημα κατά των γυναικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μικολάζικα απουσιάζει. Η κυρία Κάντεμπαχ. Όταν το 1989 εμφανίστηκε ε, το λουλούδι της ερήμου, ε, τότε ε, στο βιβλίο αυτό περιγράφεται το τι έζησε η Ροϊδά και σκέφτηκα ότι αυτό ε, θα μπορούσε να συμβεί μόνο στο Μεσαίωνα και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι συμβαίνει στην πραγματικότητα και ακόμα δεν πιστεύω ότι αυτό εξακολουθεί να γίνεται εδώ ανάμεσα μας και αφορά 500.000 γυναίκες στην Ευρώπη ε, σήμερα η κόρη μου είναι 14 ετών και είμαι χαρούμενη που δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις βάρβαρες πρακτικές νομίζω όμως ότι τώρα που γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται, καλούμεθα να διαφωτίσουμε, να ενημερώσουμε ότι δεν πρόκειται εδώ για ανθρώπινες πρακτικές, αλλά πρόκειται για κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μηδενική ανοχή. Αυτό πρέπει να ισχύει. Εδώ πρόκειται για υγεία ψυχής, ε, για ψυχική επιβάνηση. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να καταλάβουμε σήμερα είναι και να αντιμετωπιστεί ο στιγματισμός αυτών των γυναικών. Γιατί μόνο αν μιλήσουν τα θύματα ε, θα υπάρχουν και κάποιες ελπίδες να ε, δοθεί τέλος σε αυτές τις βάρβαρες πράξεις. Κύριε Κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πάρα πολλέ ακόμα οι γυναίκες και τα κορίτσια που υφίσταται αυτόν τον ακροτηριασμό. 140 εκατομμύρια υπολογίζονται και 3 εκατομμύρια κορίτσια κάθε χρόνο κινδυνεύουν. Αυτοί οι ακροτηριασμοί γενικά γίνονται σε παιδιά και φίβους από 4 μέχρι 14 χρόνια σε ε, αφρικανικές χώρες και σε βρέφη κάτω του ενός έτους. Πάρα πολλές γυναίκες ε, ε, και κορίτσια θα πρέπει τα δικαιώματά τους να γίνονται σεβαστά παντού, όχι μόνο στην Ευρώπη. Όπως είπε και ο Μάικλ Κάσμαν πριν από μένα, 500.000 είναι στην Ευρώπη γυναίκες. Είναι η σωματική υγεία αλλά και η ψυχική υγεία Κανένας λόγος, καμία πρόφαση ε, δεν δικαιολογεί αυτό. Ε, οι γυναίκες έχουν θεμελιώδες δικαίωμα να διαθέτουν το σώμα τους ίδιες. Θα πρέπει όλες οι χώρες να καταπολεμήσουν αυτή την κακομεταχείριση και ιδιαίτερα να βοηθήσουμε τις οργανώσεις που αγωνίζονται. Ε, τα είπε η κυρία Κινίλσεν και η κυρία Χιμένες Μπεσερίλ. Ευχαριστώ πολύ. Grazie. Ευχαριστώ κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Τα νούμερα είναι τρομακτικά. Δεν μπορούμε να φανταστούμε. 155 εκατομμύρια γυναικών στον κόσμο ε, θίγονται από τον ακροτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων. Θα πρέπει να φροντίσουμε εμείς στην Ευρώπη να δημιουργηθεί μια συνειδητοποίηση, να τερματιστεί αυτή η πρακτική έτσι. Θα πρέπει επιτέλους ε, να φροντίσουμε σε τρίτες χώρες να απαγορευτεί ο ακροτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων ε, οργάνων και να δημιουργηθεί συνειδητοποίηση πόσο αναξιοπρεπές και απάνθρωπο είναι αυτό. Θα πρέπει ε, τα θύματα να την χάνουν θεραπείας και ψυχικής ε, υποστήριξης για να πούμε ότι οι γονείς που κάνουν αυτό στα παιδιά τους θα πρέπει να τιμωρούνται με φυλάκιση και μάλιστα με ε, πολύ ψηλή ποινή αποτρεπτική. Ευχαριστώ. Κοστέλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ο κρατηριασμό των γενετικών οργάνων είναι και επικίνδυνο εκτός του ότι είναι αποτρόπαιο ε, ε, προσβάλλει την αξιοπρέπεια, την αναπαραγωγική υγεία των γυναικών. Πολλές γυναίκες και κορίτσια έχουν ε, ακόμα τραύματα και ουλές, όχι μόνο σωματικές και ψυχικές. Τον Απρίλιο πέρασε μια νομοθεσία και απαγορεύτηκε στην Ελλαδία και Επίσης, ε, τιμωρείται και ε, ε, η πράξη αυτή αν γίνεται εκτός Ιρλανδίας. Δηλαδή, αν φεύγουν από την Ιρλανδία πηγαίνουν κάπου αλλού και επιστρέφουν. Η Ενωμένη Νεολαία της Ιρλανδίας είναι μια οργάνωση που καταπολεμά αυτό το φαινόμενο και κάνει και επιδείξεις μόδας και άλλες δραστηριότητες. Και επίσης η Διεθνής Αμνηστία έχει ζητήσει να ε, εκπαιδεύεται το υγειονομικό προσωπικό, ιδιαίτερα στα μευτήρια, αλλά και τα σώματα ασφαλείας και οι δικαστές. Ελπίζω έτσι ε, να μπορέσει να βρεθεί και λίγη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα προγράμματα. Επίτροπε, αναφερθήκατε στην οδηγία για την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων θα έχετε ειδική αναφορά σε αυτά τα θύματα στην οδηγία, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και τέλος, Επίτροπε, καλωσορίζω πάρα πολύ το γεγονός ότι ε, δηλώσατε ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης το θέτει υπόψη και των τρίτων χωρών όταν κάνουμε εξωτερικές δράσεις. Είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτο και αυτό και σας ευχαριστώ. Grazie, Ο κύριος Ρώση. Πρόεδρε, από το 2010 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθηκε ότι θα η στρατηγική ε, περάσπιση των γυναικών και για τον γεμητικό ακροτηρισμό ε, δεν υπήρξε καμία προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. 500.000 ε, γυναίκες και παιδιά που βρίσκονται στην Ευρώπη έχουν υποστεί αυτό τον ακροτηρισμό και πάνω από 180.000 κινδυνεύουν κάθε χρόνο. Υπάρχουν κίνδυνοι υγείας και οι πρακτικές αυτές εφαρμόζονται εφαρμόζονται κυρίως σε νέα παιδιά μέχρι την ηλικία των 14 ετών στην ε, Ερυθρέα και πολλές φορές ε, και σε νεογέννητα. Ε, αυτά ε, προκαλούν πολλές φορές και τον θάνατο. Η UNICEF, η UNICEF θεωρεί τον γεννητικό ακροτηριασμό γυναικών ως παραβίαση των γυναικείων δικαιωμάτων. Εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και κατόπιν τούτου ζητώ η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει με όλα τα μέσα που διαθέτει απέναντι σε αυτές τις χώρες και να τους πει είτε θα τα δεχτείτε είτε θα καταδικαστείτε. Η κυρία Σινκλέρ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ ε, διαφωνώ ε, με αυτό το θέμα ε, σε ολόκληρο τον κόσμο υπολογίζεται ότι πάνω από 120 εκατομμύρια γυναίκες υφίστανται τον ακροτηριασμό. Ο στόχος είναι ότι η γυναίκα να είναι διαθέσιμη μόνο ε, για τον άντρα της και σε ορισμένες ε, φυλές ε, οι γυναίκες αν δεν το έχουν υποστεί δεν μπορούν και να παντρευτούν. Τα κράτη-μέλη πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα, αυτό το έγκλημα το οποίο εφόσον διαπιστώνεται στα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιβάλλονται ουσιαστικές και μεγάλες ε, ποινές. Να σταλεί ένα μήνυμα ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Ε, χάρη των εκστρατιών ε, προστασίας της υγείας έχει περιοριστεί κάπως το φαινόμενο και θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση της κοινωνίας για τις αρνητικές συνέπειες. Οι νέες γυναίκες πολλές φορές αποκλείονται για ένα ολόκληρο ολόκληρο χρονικό διάστημα. Ε, όλοι μας λοιπόν ε, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε αυτές τις βάρβαρες πράξεις. Ευχαριστούμε. Ε, το λόγο λοιπόν έχει ο Επιτρόπος κύριος Σεντάλη. Παρακαλώ. Μικρόφωνο παρακαλώ.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 Σας ευχαριστώ ε, για τη συζήτηση. Τον 21ο αιώνα εκατομμύρια γυναικών ε, υφίστανται ακόμη ε, κάθε χρόνο ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων οργάνων, κινδυνεύουν να πεθάνουν. Αν δεν επιβιώσουν μπορεί να μείνουν ανάπηρες ή να μην μπορούν να κάνουν παιδιά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί γενικότερα η βία κατά του γυναικείου φίλου και ο αγώνας κατά των ε, επιβλαβών ε, θρησκευτικών παραδόσεων όπως ο ακροτηριασμός των γεννητικών οργάνων. Ε, το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει το σχέδιο δράση για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και το στρατηγικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μία από τις προτεραιότητες είναι ακριβώς ο ακροτηριασμός των γεννητικών οργάνων. Η Επιτροπή μπόρεσε να χρηματοδοτήσει ε, έναν αριθμό, μεγάλο αριθμό προγραμμάτων της κοινωνίας των πολιτών στις ε, φτωχότερε χώρες. 50 ε, εκατομμύρια έχουν ήδη διοχετευθεί σε προγράμματα για την εκπαίδευση των νέων, για προβλήματα υγείας, για τα προβλήματα των γυναικών. Οι συνάδελφοί μου και η και Βίβια να πιστεύω ότι θα ασχοληθούν επισταμένα με την καταπολεμήση αυτού του φαινομένου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Έχουμε λοιπόν τρεις προτάσεις ψηφίσματος, καθώς έχει κλείσει η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το πρωί στις 12. Τώρα λοιπόν... Ε,